κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ολοκληρώσουμε τώρα την ε, ψηφοφορία. Απομένουν δύο εκθέσεις. Και πρώτα απ' όλα η έκθεση της κυρίας Χιάτεν Μάκη σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερβαϊτζάν. Ε, τροπολογία 2 παρακαλώ. Τροπολογία 1, με συγχωρείτε. Ε, έχουμε μια ε, προφορική τροπολογία από τον ε, κύριο Λάνμπεργκης. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για να μην υπάρξει κάποια αμφισημία, προτείνουμε μία πρόταση σε σχέση με την φράση αυτή που αφορά την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων από τον Αγκόρνο Καραμπάχ να πούμε καταρχήν να υπάρξει, at first, να υπάρξει αυτή η απόσυρση για να μην υπάρξει αμφισημία. Προφορική τροπολογία του κύριου Λάνμπεργκης. Δεν υπάρχει αντίρρηση, άρα είναι αποδεκτή η προφορική τροπολογία. Θα την θέσουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, δεν συμφωνώ με τον κύριο Λαντσμπέργκης. Λέει κυρία Μάχη εγώ υποστηρίζω το αρχικό κείμενο. βάλαμε όμως σε ψηφοφορία την πρόταση του κυρίου Λάντσμπεργκης Θα έπρεπε να υπάρχει ο αριθμός των 40 βουλευτών που αντιτίθενται. Δεν υπήρξε, οπότε η, τροπολογία, η προφορική τροπολογία τίθεται σε ψηφοφορία. Υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι κατά. Η διαδικασία αυτή διεξήχθη πριν. Ζήτησα την υποβολή ενστάσεων μετά την παρουσίαση της προφορικής τροπολογίας του κυρίου Λάμπεργκης και δεν υπήρξε ο απαραίτητος αριθμός βουλευτών. Time, Ωραία λοιπόν. Να, κάνουμε τον έλεγχο. Ακούσατε την προφορική τροπολογία του συναδέλφου Λάνμπεργκης. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ, μπορεί να υπήρξε κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της καθυστέρησης στη μετάφραση ελέγχουμε εάν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμό των 40 που δεν υπάρχει έτσι κι άλλιω. Οπότε η προφορική τροπολογία τίθεται σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ της προφορικής τροπολογίας που παρουσίασε ο κύριος Λάμπεργκης. Ήταν λιγότεροι από 40. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία... Ναι, ναι, τροπολογία 2 παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το σύνολο της πρότασης ψηφίσματος τώρα τίθεται σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Παρακαλώ, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.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 Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Πορέμπα. Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου.